Bonjour, je vous propose de, de commencer notre, notre séance. Même si je n'en ai pas le mandat, je vous prie de m'excuser au nom de la mairie de Bruxelles. Καλημέρα σας. Ε, προβλεπόταν ήλιος, αλλά τελικά δεν έχουμε. Τέλος πάντων, να θεωρήσουμε ότι είναι άνοιξη. Ε, η Μαρίτα δεν μπορεί να έρθει δυστυχώς, γιατί τώρα διεξάγεται η σε κοινωνική ε, σύνοδος ε, και δεν θα μπορέσει να έρθει. Έχουμε διερμηνία για όλες τις γλώσσες εκτός από τα κροατικά. Για τα πρακτικά τώρα που συνεδριάζει 21 και 22 Φεβρουαρίου, 26 και 27 Φεβρουαρίου τα έχετε δει και δεν ε, υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Θα δώσω το λόγο στην Ανιές και στην Ελίζαμπέτ αμέσως. Του είχαν πολύ φορτωμένες βραδιές από ό,τι κατάλαβα. Δεν νομίζω να κοιμηθήκανε και πολύ. Είσαστε στον 8ο τριμερή διάλογο, αν δεν κάνω λάθος. Ε. Θα σας δώσω το λόγο συνοπτικά, αν μπορείτε να μας πείτε τι έχει γίνει Ε, κυρία Μωρά Σατιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε και θα, θα αρχίσω εγώ και όπως συνηθίζουμε θα συμπληρώσει η Ανιές. Ο 8ος τριμερής διάλογος. Τι έχει γίνει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Να με διορθώσει ο Ρομπέρ άμα ε, κάνω κάποιο λάθος γιατί ήταν μαζί μας. Πρώτον, ε, καταλήξαμε σε μια συνολική συλλογική συμφωνία για το διατακτικό. Ε, δουλέψαμε τα άρθρα μαζί με το Συμβούλιο. Αυτό έγινε ε, πριν από ένα δεκαπενθήμερο και μετά τη Δευτέρα το βράδυ αποκρισταλώθηκε αυτή η συμφωνία ανά άρθρο και μετά περάσαμε σε τελική σκέψη, τα εκτιμώντας. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί στις 9 παρατέταρτο, αγαπητή μου Άγνες, νομίζω μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τις ε, διαπραγματεύσεις, ε, δηλαδή ε, αποκρισταλώθηκε η συμφωνία μέσα, και το λέω αυτό διότι διεξοδικά εξετάσαμε όλα τα άρθρα του διατακτικού και έκλεισε, κλείδωσε η συμφωνία. Όταν είναι έτοιμα τα έγγραφα θα σας τα στείλουμε. Τι γίνεται τώρα με τις διαπραγματεύσεις και την έκβασή τους. Χρονικά, ας δούμε τη, τη χρονική κλίμακα γιατί και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. καταλήξαμε ε, σε συμφωνία για την κοινοποίηση προς το κράτος μέλος υποδοχή από πλευρά της επιχείρησης σε 12 μήνες συν 6. Δεύτερο σημαντικό σημείο ήταν στη διαπραγματευτική μας εντολή, θα το θυμάστε. Έχουμε διτή νομική βάση κατοχυρώντας έτσι ταυτόχρονα την προστασία των εργαζομένων και την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για την εγχώρια αγορά μέσα στην ε, οδηγία. Εγώ τώρα σχεδιαγραφώ γενικές γραμμές, η Αγνία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Διευρύνουμε την οδηγία του 96, δεν είναι νέα η νομική βάση. Προβλέπεται μέσα σε ένα άρθρο το Συμβούλιο ήθελε να μπει σε αιτιολογική σκέψη. Όμω ε, ε, οι διαπραγματεύτριες ήταν ιδιαίτερα επίμονες ε, και τα καταφέραμε τελικά. Επιβληθήκαμε και η νομική βάση συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο και αυτό θα είναι σημείο αναφοράς σε σχέση με την μελλοντική νομολογία του ΔΕΚ. είναι στο πρώτο άρθρο. Για την αμοιβή Έμειναμε στη κοινή μας θέση, δηλαδή πρόκειται για τον ελάχιστο μισθό του κράτους υποδοχής και τα μπόνους που συνδέονται με το μισθό, ούτως ώστε μισθολογικά να εξισώνονται οι ε, εργαζόμενοι του κράτους ε, υποδοχής και οι αποσπασμένοι. Η εργασία, ίσως μισθός λοιπόν για τον ίδιο χώρο εργασίας. Για τις ε, αποζημιώσεις, λάβαμε υπόψη διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν ανάλογα με τη χώρα. Μπορεί να καταληφθούν οι αποζημιώσεις από τη χώρα προέλευση ή τη χώρα υποδοχής και ούτω καθεξής. φροντίσαμε το gross amount, το ακαθάριστο ποστό, να είναι ίδιο για τους εργαζομένους της χώρας πρέλευσης και χώρας υποδοχής. Για τις ε, συλλογικές ε, συμβάσεις ε, θα μας δώσει λεπτομέρειες οι Ανιέζε. Μόνο επιτρέψτε μου να σας ε, να αναφερθώ σε δύο σημεία όπου αγωνιστήκαμε με νύχια και με δόντια για τη μεταβατική περίοδο και για την προθεσμία εφαρμογής. Θυμάστε στο κείμενο του Συμβουλίου είχαμε τριετή μεταβατική περίοδο για κανένα κράτος μέλος δεν μπορούσε να μεταφέρει στην Εθνική Νομοθεσία πριν να εκπνεύσει αυτή η περίοδος των ε, τριών ετών και η περίοδος εφαρμογής ήταν τέσσερα χρόνια. Για μένα ήταν ιδιαίτερο σημαντικό να γίνει πλήρω σεβαστή η διαπραγματευτική μα εντολή. Δύο χρόνια μεταβατική περίοδο, δύο χρόνια ε, περίοδος εφαρμογής για να ε, σεβαστούμε και την νομοτεχνική εργασία του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δέχτηκε το Συμβούλιο. Δύο συν δύο λοιπόν. Τέλος. Καταφέραμε να διορθώσουμε ένα σημείο που ήταν ιδιαίτερο σημαντικό για τους ε, Ισπανούς και Πορτογάλους ε, συναδέλφους για τη μεταφορά. Λέει, δεδομένης δουλειάς που γίνεται για το Lex Specialis. Η μη τροποποιημένη οδηγία του 96 θα είναι εφαρμοστέα μέχρι την εφαρμογή της ε, ειδικής νομοθεσίας. Το Συμβούλιο και διαπράξει ένα μικρό λάθος τον Οκτώβρη. Είχε μιλήσει για την θέση σε ισχύ. Ότι θα ίσχυε η οδηγία των 96 μέχρι θέση σε ισχύ του Lex Specialis, όμως αυτό δεν ισχύει γιατί η θέση σε ισχύ είναι πρώτερη της ε, θέσης εφαρμογή. Θα χρειαζόμασταν τρία καθεστώτα 96 μέχρι να τεθεί σε ισχύ, η, 96, η διοδηγία, η του 96 ε, για την περίοδο από θέση ισχύ μέχρι τη θέση εφαρμογή και μετά λέξη specialis. Πολύ δύσκολο ήταν για τα κράτη-μέλη να αλλάξουν καθεστώς τρεις φορές. Δέχτηκε το Συμβούλιο λοιπόν η θέση σε εφαρμογή να είναι ε, αυτό που σηματοδοτεί τη εφαρμογή του Lex Specialis. Θέλω να πω πως δύσκολα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις για τόσο περίπλοκο κείμενο που, όπου υπάρχουν τόσο διαφορετικά συμφέροντα. Πάντως ε, με τις προσπάθειές μας υπήρχε ισορροπία ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση της Ευρώπης μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη τα αιτήματα των ΜΕΝ και των ΔΕ και καταφέραμε να μην υπάρξει ρήξη και χάσματα. Καταφέραμε Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ε, προστασία των εργαζομένων και το σεβασμό των επιχειρήσεων, ε, των συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά. Τα καταφέραμε να τα ενσωματώσουμε στο κείμενο, Εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και όταν ε, τα βάλαμε με το Συμβούλιο και είχαμε αυτή τη διελκυστίνδα, τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά και πέρασαν τα βασικά σημεία του Κοινοβουλίου. Σε ευχαριστώ θερμά, ε, Ανιές, για τη συνεργασία μας. Σπανίζει, ξέρετε, δύο συνεισηγητές από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, να συνεργάζονται με ειλικρίνεια και ενωμένη. Όμως επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, σκιώδεις ε, συγκριτές που ακολούθησαν την όλη διαδικασία με ιδιαίτερη προσήλωση και μας ζητούσαν να κάνουμε και διακοπές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ούτω ώστε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να εξασφαλίζουμε κάθε φορά την σύμφωνη γνώμη των σκιωδών. Πολύ καλή ομάδα μας και δεν εννοώ μόνο την Ανιές ε, και εμένα, αλλά και τους ε, συναδέλφους, ε, τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία αυτό ο ακρογωνίος λήθος της κοινωνικής Ευρώπης εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you, Chair, and... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που, κατασ δυνατό, εφικτό να ε, φτάσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό, σημαντική φάση την περασμένη Δευτέρα. Και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει την Ελίζαμπεθ και τους Κιώδης, καθώς και την ε, Γραμματεία. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμο το έργο της ε, νομικής υπηρεσίας και όλων των βοηθών. Γιατί αυτή τη στιγμή αναπόκειται σε εμάς τους ε, δυο μας, αλλά και τους ε, Σκιώδης και την Βουλγαρική Προεδρία να ε, κερδίσει την υποστήριξη για τις συμφωνίες που έγιναν την περασμένη Δευτέρα. Και εάν κατάλαβα καλά, έχουν, σήμερα υπάρχει, θα γίνει μια ενημέρωση με το Κορεπέρ και θα ακολουθήσει μια επιστολή την οποία θα λάβουμε εμείς μετά από τη συνεδρία του Κορεπέρ στις 11 Απριλίου. Και στη συνέχεια θα κάνουμε τα τελευταία βήματα που είναι αναγκαία. Έμαθα πολλά πράγματα από όλη αυτή τη διαδικασία και Νομίζω ότι κάναμε πραγματικά κάτι που έχει μια αξία για τους Ευρωπαίους εργαζομένους και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι. Όπως είπε η Ελίζα Μπέθε, κάναμε κάποιες ε, αλλαγές ε, στις πολιτικές συμφωνίες που έγιναν πριν από δύο εβδομάδες για τα επιδόματα Επίσης, προκειμένου να κερδίσουμε την υποστήριξη του Συμβολίου από την Τσεχία και τη Σλοβακία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί αυτή η συμφωνία χρειάζεται μια πλατιά υποστήριξη και γι' αυτό δεν επιμείναμε σε κάθε ε, μέρους διατύπωση. Αλλά προσπαθήσαμε τη Δευτέρα να προσαρμόσουμε και να καθισχάσουμε τις, ε, το κείμενο να καθισχάσουμε τις ανησυχίες των διαφόρων χωρών ε, μελών και να υπάρξει μια νομική σαφήνεια όσον αφορά τις ε, αποζημιώσεις για τα έξοδα ταξιδίου κλπ. Και, και διορθώθηκαν κάποια σφάλματα τα οποία είχαν γίνει πραγματικά στο Συμβούλιο ε, όσον αφορά τις ε, εξαιρέσεις σε σχέση με τις μεταφορές και ήταν σημαντικό να κερδίσουμε την υποστήριξη των Πορτογάλων και θα ήθελα επίση να ξεκαθαρίσω ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές ε, έχουν μια νομική κατοχήρωση μέχρι να ισχύσει το ΛΕΚ Σπεσιάλης e γιατί συνεχίζει να ισχύει η προηγουμένη νομοθεσία και υπολογίζουμε στη στήριξη των χωρών μελών για την ενδιάμεση περίοδο προκειμένου να εφαρμόσουν τον κανονισμό που υπάρχει από το 1996. Και κατόπιν ετήματος των ε, Σουηδών ε, διαφερομένων ε, ξεκαθαρίσαμε κάπως <clears throat> τη διατύπωση σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να καταστήσουμε το σαφές <clears throat> ότι μιλάμε ακριβώς για συλλογικές διαπραγματεύσεις και εδώ ε, είναι οι χώρες μέλη που θα δηλώσουν την καθολική τους εφαρμοσιμότητα, διευρύνοντας την εφαρμαγή, εφόσον το επιθυμούν, όχι μόνο αυτές που ισχύουν καθολικά, είναι καθολικά εφαρμοστές, αλλά και τις ε, ε τομεακές ε, συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις. Επίσης ξεκαθαρίσαμε ότι αν ε, στις χώρες μέλη, όπως ισχύει στις ε, σκανδιναβικές χώρες, δεν είναι κυβερνήσεις αλλά κοινωνικοί εταίροι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και αυτό είναι εντάξει και καλύπτεται από το άρθρο αυτό. Επίσης κάναμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις υπεργολαβίες όπου ξεκαθαρίσαμε ότι στην ιδιολογική σκέψη αναφερόμαστε στην οδηγία εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς ε, κανόνες όσον αφορά την ευθύνη στις ε, υπεργολαβίες και Συνολικά θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα πολύ τεράστιο βήμα προς τα μπρος, γιατί είναι πολύ βασική η αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία στο χώρο εργασίας και αποτελεί και ένα βήμα προς τα μπρος, γιατί όπως είπε ήδη η Ελίζαμπεθ, ε, νομίζω ότι βαθμιδών ε, μπορέσαμε να εξορροπήσουμε τα, τα συμφέροντα εργαζομένων και εργοδοσίας στις διάφορες χώρες μέλη και διαφόρων ε, ομάδων συμφερόντων και επίσης πετύχαμε κάποιες πρόοδους μέσω της θέσπισης ξεκάθαρων και εφαρμοστέων κανόνων <clears throat> και ίσως σε μια ε, προσεχή φάση, ίσως το Μάιο, θα έχουμε εδώ μια ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, αφού το κείμενο <clears throat> έχει αποσταλεί μέσω επιστολής από την Κορεπέρ, αλλά θα αξιοποιήσω και το διάμεσο διάστημα μέχρι την ψηφοφορία, ούτε ώστε να πείσω όσο δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να το υπερψηφίσουν, γιατί πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις στην Ευρώπη ε, πραγματικά μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις πρόοδου. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία που έγινε είναι ξεκάθαρο ότι μεν και οι δε θα πρέπει να τοποθετηθούν ε, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο σε συνάρτηση με το τελικό κείμενο και φαντάζομαι πως ότι και οι δύο είστε σε θέση, στη διάθεση των ενδιαφερόμενων προκειμένου να κάνετε κάποιες διευκρινήσεις και να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες και αυτό θα περάσει στην Ολομέλεια, θα ψηφιστεί τον Ιούνιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Αρκετά σημαντικό αυτό όσον αφορά την ε, πρόθεση της υπόθεσης απασχόλησης. Ο κύριος ε, Μητροφάνος είναι ο εισηγητής. Sorry. Oui, ένα ερώτημα στους συνεισηγητές, λέει ο κύριος Καλβέ Σαμπών. Όχι, όχι, να γίνει συζήτηση. Θέλω τη συζήτηση. Αλλά αν ανοίξουμε τώρα συζήτηση και όλοι λάβουν το λόγο, τότε με τα δεδομένα χρονικά πλαίσια δεν θα βρούμε άκρη. Όμως, όμως, για να επαναλάβω το οποίο είπατε, είμαι στην ε, διάθεση όλων, οπότε μπορούμε να τα πούμε είτε σε επίπεδο πολιτικών ομάδων, είτε αντιπροσωπιών, είτε ε, διμερός προσωπικά, λέει η κυρία Μόνα Σατιέ. Για αυτό το το που θέλατε. Κύριε Μητροφάνος. Uh, uh, uh, πρώτα πρώτα συνάδελφοι θα πρέπει να σας πω κάποια τεχνικά σημεία. Αν μια ματιά στη βάση του του κοινοβουλίου. Θα δείτε τα σχετικά με αυτές τις κατευθυντήριες για τις ε, πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ε, και έχουμε τις τροπολίες κυρίας Ντανόκα. Ε, εγώ την αντικατέστησα όταν απεχώρησα από το κοινό πριν από ε, τρεις εβδομάδες και οπότε μου κληροδότησε αυτή τη ε, δουλειά και να ευχαριστήσω επομένως πρώτα πρώτα όλους τους χιώδεις εισηγητές γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, παραγωγική η δημιουργική συζήτηση χτες που τα είπαμε και προσπαθήσαμε πραγματικά να λάβουμε υπόψη όλα όσα ε, είπαν και ήθελαν οι συνάδελφοι οι περισσότεροι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη έκθεση. Είναι ειδική περίπτωση μια που πριν από δύο εβδομάδες το Συμβούλιο, η Βουλγαρική Προεδρία συγκεκριμένα μας είπε ότι όταν το Κοινοβούλιο ψηφίσει αυτή την έκθεση θα ληφθεί, ίσως θα ληφθεί τέλος πάντων υπόψη από το Συμβούλιο ένα, ένα βήμα πρόοδου και για την Επιτροπή μας και για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Τι θα γίνει τώρα τις αμέσως εβδομάδες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την διαδικασία έγκρισης της έκθεσης. Χθες καταλήξαμε σε κάποιες πολύ θετικές συμβαστικές τροπολογίες. το έγγραφο το στείλαμε σε όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές κατά το βραδάκι. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε την έκθεση για ψήφιση στην ε, Σύνοδο του Μαΐου, αλλά να δούμε τι εξυπηρετεί καλύτερα. Σαν λέγαμε για 25 ή 26 Απριλίου. Όμως, Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 27 Μαρτίου. Ε, βέβαια και ακούσαμε τις παρατηρήσεις όλων των στέλνων από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα λάβουμε όλα όσα είπαν υπόψη. Και νομίζω ότι θα είναι λίγες οι τροπολογίες που θα κατέβουν προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Γιατί όπως σας είπα κάναμε ό,τι μπορούσαμε ε, περισσότερο για να μπορέσουμε να κλείσουμε και συμβασμούς ε, με τους χιώδης ηγητές. Τώρα, για το ΕΛΚ, ο κύριος Πλούρα. Έχεις. Σας ευχαριστώ. Όπως είπαμε ε, χθε στη σύσκεψη των σκιωθών εισηγητών, εισηγήθηκε ο κ. Μητροφανού να επιτεχύνουμε την ε, εργασία μας και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις για τις ε, τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μητροφάνους που δέχτηκε να συνεχίσει την δουλειά της συναδέλφου. Ε, κατάφερε να εκπονήσει ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι συμπληρώνουν πολύ καλά το έγγραφο οι τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Και χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που ελέγξαν υπόψη αυτές οι τροπολογίες. Η νέα εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών ανταποκρίνεται ε, πλήρως ε, στις συζητήσεις που έγιναν στο πρώτο γύρο. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Ε, χαιρόμαστε που ε, λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα των μικροεπιχειρήσεων και των μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως είπε όμως και ο συνάδελφος Ανταμκός, Ε, θα πρέπει πάντοτε να συνεχίσονται οι κοινωνικές διαπραγματεύσεις, ε, γιατί πολλές φορές συμβαίνει ε, να συμβαίνουν, να, να διεξάγονται με μεγάλη καθυστέρηση και τελικά ε, σε σχέση με την τροπολογία 18 πρέπει να πω ότι θα πρέπει να δρούμε εγκαίρως ως προς διαπραγματεύσεις. Τώρα για τους κοινωνικούς εταίρους Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί διαφορετικοί και θα πρέπει να καλυφθούν όλοι. Επίσης, τροπολογία 5, μην ξεχνάμε το σύμφωνο σταθερότητας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όργανο της οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί μίλησαν για τη συμφιλίωση οικονομικής και επαγγελματικής ζωής, Θέλω λοιπόν να πω πως ε, είναι ε, καλές όλες αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας ε, και για τους εργοδότες και για τους εργαζομένους. Θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία και στο Συμβούλιο και κυρίως θα επιμείνουμε ώστε να ληφθούν υπόψη τα σημαντικά για το Κοινοβούλιο σημείο. Ελπίζουμε να καταλήξουμε συνετική λύση μέχρι το τέλος της τρέχουσας ε, εβδομάδας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 27. Ε, Εάν δεν τα καταφέρουμε, προτείνω να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής του Στρασβούργου. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ντέτχεν, για τους σοσιαλδημοκράτες. Το μικρόφωνο του δεν έχει ανοίξει. Sorry. I start again. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μητροφάνος ε, για την ε, δουλειά που έκανε για να συνεχίσει τη δουλειά της κυρίας Αουτνόγκα. Εργάστηκε ταχύτατα και αποτελεσματικά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θετικά μηνύματα που μας πέρασε το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις και φυσικά θα εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία και από πλευράς μας, ούτως ώστε ε, ταχύτατα να διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα. Όσο ταχύτερα εγκριθεί ε, το σχέδιο, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και την κατάσταση επιτόπου μέσα από το, το νέο αυτό όργανο. Α, για αύριο έχουμε προγραμματίσει και άλλη σύσκεψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, εγκριθούν και οι 20 αρχές ε, της κοινωνικής Ευρώπης. Ε, φυσικά θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφερθούμε στην εγγύηση για τους νέους, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν πολύ καλές ευκαιρίες οι νέοι. Μέσα στην έκθεση καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις στις πολιτικές ομάδες και ε, είναι αρκετά ε, σταθερή η έκθεση, αλλά όμως χρειαζόμαστε και ε, διευκρινήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές, παραδείγματος χάρη για τη συνταξιοδοτική πολιτική, για τα κράτη-μέλη, για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα και χρειαζόμαστε σαφήνεια. Δηλαδή να καλύπτουμε όλη την, όλο το φάσμα από τους νέους μέχρι τους συνταξιούχους. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε διευκρινήσεις για κάποια υποσημεία. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κανένα από τους φιλελεύθερους, ούτε από την ΚΟΕ. Η Λάουρα Συνάδελφοι, ευχαριστούμε ε, και μπράβο που κλείσαν αυτούς τους ε, συνδεσμούς. Μου φαίνεται ε, ότι είναι δημοκρατικό αυτό το οποίο διαμορφώνει τα τελευταία χρόνια γιατί τελικά είναι ένα στεγανό έγγραφο που βγήκε από τις επιτροπές μας και ανέκαθεν δεν τα λάμβανε αυτά υπόψη το Συμβούλιο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αυτή η φάση παρακάμφθηκε, ξεπεράστηκε και άρα θα ολοκληρώσουμε έτσι αυτήν την ε, πρόταση και αυτό θα αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία περιμένουν ε, οι πολιτούς τους οποίους και το κοινοβούλιο τους ε, εκπροσωπεί και έτσι θα ακουστεί δυνατά η φωνή τους οπότε θα πρέπει όσο γίνεται πιο σύντομα να συμφωνήσουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας ή να καταστεί ο στόχος μας τώρα όσον αφορά τις προτεραιότητές μας. Ε, είδαμε τι έγινε τελευταία διετία. Εγώ ήμουν η, η και θα τις έχω αναδείξει αυτές τις προτεραιότητες το ώστε να δούμε το ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια σε κάθε μορφή της σήμερα στην Ευρώπη. Γινόμαστε μάρτυρες ενισχυτικού φαινομένου, δηλαδή τους φτωχούς εργαζόμενους. Είναι αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν δουλειά αλλά κινδυνεύουν να πέσουν σε φτώχεια και τα νούμερα όλο ένα και φουσκώνουν. Έχουμε ταυτόχρονα και τις ευάλωτες ε, θέσεις ε, εργασίας, άρα στόχος μας είναι να υπάρχει ε, βέβαιη δουλειά και αξιοπρεπής. Επομένως, θα πρέπει να αλλάξει η στάση των κρατών μέλων. Όμως υπάρχουν ε, ε, οι δημοσιονομικοί κανόνες, τα δημοσιονομικά σύμφωνα, ε, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας και τα κρατη δεν είναι ελεύθερα να θεσπίσουν, να, να δημιουργήσουν τέλος πάντων θέσεις ε, εργασίας ποιοτικέ. Προσοχή γιατί θα υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να φρενάρουμε την φτώχεια και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων. Επίσης θα πρέπει να μην έχουμε ιδιαίτερο φορολογικό βάρος προς τις ΜΜΕ ή και γραφειοκρατίας βάρος τους. Γιατί εκεί δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και άρα αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι στη θέση να το κάνουν. Επίσης ε, θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τη φορολόγηση της εργασίας, να προσέξουμε όσον αφορά τις βιώσιμες ε, πηγές ενέργειας και να δούμε τι θα κάνουμε τα ορυκτά καύσιμα. Να βρούμε δηλαδή, να δώσουμε κάποια λύση στο ενεργειακό που να βοηθά τις ΜΜΕ. Και υπάρχει ένα άλλο σημαντικό θέμα. Αφορά τους νέους και τους μακροχρόνιους άνεργους. Για τους ε, νέους. Θα πρέπει να τους ε, καταρτίζουμε, να έχουν δεξιότητες, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διορθωτικές αλλαγές της δουλειάς και επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά που ξέρουν τις δεξιότητές τους μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και να μπορούμε να τους εντάξουμε στους νέους κλάδους, στις νέες δουλειές που δημιουργούνται από την πράσινη, την κυκλική, την μπλε οικονομία. Ε, προς τα εκεί να τους καταρτήσουμε. Οπότε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις ε, αλλαγές που τώρα αναδύονται, που είναι έντονες και αφορούν το μετασχηματισμό της δουλειάς. Να δούμε επίσης ε, πώς θα διαχειριστούμε τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση, όλα αυτά πρέπει να τύχουν της προσοχής μας να σταματήσουν οι δυσμενείς διακρίσεις, και να υπάρχει συγκερασμός ιδιωτικού βίου και επαγγελματικού βίου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει, λέω, να το προσέξουμε, να είμαστε αποφασιστικοί. Γιατί μπροστά μας έχουμε σημαντικές αλλαγές της κοινωνίας. Άρα, να συνδυάζονται, να συγκεράζονται ε, αυτά τα δύο και να υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας χωρίς να έχουμε στρεβλώσεις, να υπάρχουν εγγυήσεις για κοινωνικές ε, υπηρεσίες όπως εκπαίδευση παιδεία των παιδιών κλπ. Να είναι επομένω ρωμαλαίο το κοινωνικό σύστημα και ο ιδιωτικός και κοινωνικός βίος να συνδυάζεται με τον επαγγελματικό. Επίσης να βοηθήσουμε τις νέες μορφές εργασίας, smart working, τηλεεργασία. Να υπάρχουν εγγυήσεις και να μην έχουμε με αυτές τις νέες μορφές εργασίας καταχρήσεις και παράκαμψη του νόμου. Να μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι να υλοποιούν το, τα, τα σχέδιά τους σε επίπεδο επαγγελματικό τελευταίο και ας είναι σημαντικό είναι το θέμα των συντάξεων στόχος μας είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα που αυξάνεται το συνταξιοδοτικό ηλικιακό όριο. Συνέχεια αυξάνεται. Όμως αυτό δεν είναι βιώσιμη απάντηση στα προβλήματα. Θα πρέπει βέβαια να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να επιλέξουν, να ξέρουν τι προοπτικές απασχόλησης έχουν, να γίνεται η αναλλαγή των ε, γενεών να γίνεται ε, αλλαγή σκητάλης όσον αφορά τις ε, δεξιότητες μέσα στις ε, αλλαγές που αναδύονται στα κρατή-μέλη, στην Ευρώπη γενικότερα και να βρεθεί έτσι η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Να δούμε τι θα γίνει με το συνδεξιωτικό ηλικιακό όριο και πώς θα καλύψουμε τους εργαζόμενους που είναι σε ευάλωτες θέσεις εργασίας να μην υφίστανται την σημερινή εκμετάλλευση. Ε, ναι, τα, τα όσα είπε η κυρία Σεά, εγώ θα είμαι ε, πολύ πιο σύντομο γιατί ήδη έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις και ε, υπάρχουν και έχουν τα 14 τροπολογίες που ελπίζω ότι θα τις υπερψηφίσετε. Είναι ένα θέμα το οποίο το ξαναβρίσκουμε κάθε χρόνο, σχεδόν με την ίδια διατύπωση, με τους ίδιους ευσεβείς πόθους, τα ίδια εργαλεία ε, και ε, τελικά τις ίδιες ε, παρακάμπτηρίους για να καταλήξουμε στο σημείο αυτό. Ε, ε, γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός γιατί μπορώ να προδικάσω ότι τα αποτελέσματα θα, δεν θα είναι θετικά, θα είναι αρνητικά. Ε, νομίζω ότι ήμουν αρκετά σύντομος. Ε, ναι, βεβαίως λέει ο Πρόεδρος. Ε, κυρία Σέστομα από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης έχει το λόγο. <coughs> Α, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που δώσατε το λόγο στην Επιτροπή. Ε, χαιρετίζουμε τις ε, πάνω από 100 τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί και θα ελπίζουμε να διεξαχθεί η ψηφοφορία την προσεχή εβδομάδα και θα δούμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. πράγματι, ε, είχαμε προγραμματίσει την 25η-26η Απριλίου. Ε, ίσως θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα και για να πάει συνέχεια στην Ολομέλεια το Μάιο. Τώρα θα περάσω στο επόμενο σημείο που αφορά ε, ε, την παρουσίαση μελέτης για τα βοηθητικά εργαλεία για τα άτομα με αναπηρία. Ε, πρόκειται για σημαντικές ε, μελέτες και θα δώσω αμέσως ε, το λόγο στον κύριο Άνταμ Κοζά για δύο ή τρία λεπτά, αν το επιθυμεί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή μας ε, ασχολείται με σημαντικά θέματα για τους ανθρώπους με αναπηρίες και το 2015 ε, προτείναμε η ΣΤΟΑ να εκπονήσει μια επιστημονική μελέτη. Πώς ε, λειτουργούν αυτές οι βοηθητικές τεχνολογίες για την καλύτερη ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες. Ε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, νοητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω αυτών των νέων τεχνολογιών. Γιατί αυτές οι τεχνολογίες ε, μελλοντικά θα έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινή μας ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το πώς θα πειράσουν τεχνολογίες αυτές στη ζωή μας με ποιες ε, επιπτώσεις ε, ε, και τι είδους επιπτώσεις θα έχουν εφόσον διαδοθούν. Ποια θα είναι δηλαδή η βιώσιμη επίδραση των τεχνολογιών αυτών στις κοινωνίες μας. Και εν μέρη χωρίς να υπάρχει αυτή η πρόθεση εκ των προτέρων πρέπει να δούμε εμείς από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς τοποθετούμεθα έναντι αυτών των τεχνολογιών. Βεβαίω, υπό την προπόθεση θα λάβουμε υπόψη μας ε, την, Ευρωπαϊκή Χάρτα και θα διευρύνοντας την ε, άρση των φραγμών. Υπάρχει λοιπόν ένα ιατρικό πρίσμα και το πρίσμα των ε, εργαζομένων. Σημαντικό εδώ είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά αυτά τα βοηθήματα και να λάβουμε αποφάσεις ε, γνωρίζοντας το μέγεθος της ευθύνης μας. Υπάρχουν και κοινωνικά, ηθικά, νοητολογικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Γιατί ε, η τεχνολογία κάνει άλματα, αναπτύσσεται ραγδαία. Ε, φοβόμαστε ότι η νομοθετική μας ε, ταχύτητα ή μάλλον βραδίτιδα ε, μένει πίσω από την πραγματική ζωή. Εγώ περιμένω με ανυπομονησία την σύναψη των εμπειρογνώμων που εκπώνησαν την μελέτη και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να διαβάσουν την μελέτη και η βοηθή γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάγια, η οποία έκανε μία κολοσιαία μελέτη, ποσοτικά, από ποσοτική άποψη, αλλά ε, έχει τη διάθεσή της 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια ανάλυση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση και την ε, μελλοντική διαμόρφωση των τεχνολογιών αυτών. Ε, προσεχήσαμε τρεις ε, αναπηρίες, ε, οπτική, ε, ακουστική και ανθρώπους που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Δώσα, επικεντρωθήκαμε στο θέμα της κοινωνίας, της κατάρτισης και των θέσεων απασχόλησης. Θα αναφερθώ τώρα και θα αναφερθώ σήμερα στο θέμα της ε, απασχόλησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος ε, καταρτήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ε, διανύμαμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες εάν χρησιμοποιούν κάποιο, κάποιο βοήθημα για να βελτιώσουν την αναπηρία τους και είδαμε ότι οι απαντήσεις ήταν θετικές. Επίσης, τους ρωτήσαμε ειδικά σε ποιο τομέα τεχνολογίες αυτές ήταν σημαντικές όσον αφορά την παροχή υποστήριξης. Και όπως μπορείτε να δείτε στις ε, διαφάνειες τις οποίες ε, παρουσιάζω, ε, κάθε μία επικεντρώνεται στο είδος της αναπηρίας και διαπιστώνουμε ότι το σχολείο και η εργασία είναι οι βασικοί τόποι που χρειάζονται τέτοιου είδους υποστηρικτικές ε, τεχνολογίες υποστηρίζοντας ανθρώπους με αναπηρίες και δυσκολίες ιδιαίτερα στον τομέα της ε, εκπαίδευσης αλλά και της εργασίας. Επίσης ζητήσαμε να μας δώσουν κάποια παραδείγματα τέτοιου είδους τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τόπο εργασίας. Και βεβαίως οι απαντήσεις ε, σύμφωνα ήταν σύμφωνα με τον τύπο, ανάλογες με τον τύπο της αναπηρίας και περιλάμβαναν ιατρικές συσκευές αλλά επίσης και τεχνολογίες mainstream. Για παράδειγμα, ε, τεχνολογίες πληροφορικής και εφαρμογές, δηλαδή ε, μεγεθυντικές ε, οθόνες ή ήταν χρήσιμες για τους τυφλούς ή τα, άτομα με προβλήματα όρασης. Επίσης, τεχνολογίες ε, ε, σε κείμενα ή ε, τεχνολογίες πληροφορικής που μετατρέπουν ε, οπτικά κείμενα σε ηχητικά σήματα. Επίσης δόθηκαν παραδείγματα και για τους τρεις τύπους αναπηριών. Για παράδειγμα, η μεγέθυνση ε, προβολή της πραγματικότητας στην περίπτωση του αυτισμού για να υποστηριχθούν οι κοινωνικές αλλαπιδράσεις στο χώρο εργασίας και για παράδειγμα με παιχνίδια μπορεί να πάει κανείς στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να πει καλημέρα στους συναδέλφους και γίνεται μια προσωμο... προσωμείωση των συναδέλφων γιατί η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι δύσκολη για άτομα με... που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό το οποίο θέλαμε είναι να υπάρχει μια λογική προσαρμογή για τα άτομα με αναπηρίες και αυτό ε, αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος για την εκπόνηση αυτών των ε, τεχνολογιών υπάρχουν εύκολες προσαρμογές που μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η ένταξη των αυτιστικών ατόμων στο χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν δούμε τον αυτισμό, τα κοινωνικά μέτρα ή η, ε, ε, η, συμπεριληψη ενός βοηθού στο χώρο εργασίας μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, επειδή τα αυτιστικά άτομα είναι υπερβέσθητα σε ήχους και στο φωτισμό, ε, θα, ε, είναι δυνα... θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος εργασίας όπου να αμβλύνονται αυτά τα ρεθίσματα, τα οπτικά και τα ηχητικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διακρίσεις σε σχέση με τους ε, ανθρώπους με αναπηρία ήδη στη φάση της πρόσληψης. Επίσης υπάρχουν ε, έλλειψη, δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση ε, όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την εργοδοσία. Η εργοδοσία τελικά εξετάζει το, το φορτίο και το κόστος και προκειμένου να προσλάβουν ανθρώπους με αναπηρία και δεν εφαρμόζονται καθόλου και οι κυρώσει στην περίπτωση που επιχειρήσει αρνούνται να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες. Άρα λοιπόν και υπάρχει μια γενική έλλειψη γνώσεων όσον αφορά ανθρώπους με αναπηρίες ε, σε σχέση με το χώρο εργασίας. Επίσης υπάρχουν ελλείμματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί μια καλή εκπαίδευση θεωρείται προϋπόθεση για ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, όπως είδαμε από τη μελέτη, εάν άτομα με αναπηρίες δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ε, λόγω των ελλείψεων προσαρμογών όσον αφορά ε, και τις τεχνολογίες, το τελικό αποτέλεσμα είναι ε, άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και χαμηλές δεξιότητες θα έχουν δυσκολίες να βρουν ε, εργασία. Όχι λόγω της αναπηρίας, αλλά κυρίως λόγω του χαμηλού επίπεδου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να ευσύσω την προσοχή στα εξή ε, θέματα. Το ένα είναι η σημασία τελικά να εφαρμοστεί η σύμβαση να διασφαλίσουμε ότι έχει μεταφερθεί στον κανονισμό της κάθε χώρας και θα πρέπει να επιβληθούν, να αξιολογηθεί η εφαρμογή και να επιβληθούν κυρώσεις στις χώρες που δεν συμμορφώνονται. Επίσης ε, θα πρέπει οι τεχνολογικές ε, ε, δυνατότητες να συνδεθούν με την κοινωνική σφαίρα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του χρήστη η μελλοντική εξέλιξη των τεχνολογιών δεν θα πρέπει να εξετάζει μόνο τις νέες συσκευέ, αλλά και την ε, δυνατότητα βελτιωμένης εφαρμογής των ήδη υφιστάμενων. Αυτό ε, Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια εξολόγηση των ήδη υφιστάμενων εφαρμογών και να υπάρξει μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών. Επίση, όσον αφορά την ίσχυση τη εκπαίδευση, η γνώση για το πώς να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προκειμένου να ε, υπάρξει μια βελτίωση, ε, θεωρείται ως σημαντικός παράγον για την απασχολησιμότητα ανθρώπων με αναπηρίες. Δηλαδή θα πρέπει να καταρτιστούν τουν τα άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τη χρήση και τον ρόλο αυτών των βοηθητικών μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να καταρτιστούν και οι επαγγελματίες στις δημόσιες υπηρεσίες, οι μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες της υγείας, αστυνομικές δυνάμεις κλπ. Και ε, θα πρέπει να ε, ξέρουν πώς μπορούν να προσεγγίσουν ένα άτομο με αναπηρίες και πώς μπορούν να παράσχουν υποστήριξη. Ε, και με αυτό συνδέεται η ανάδυση ενός ε, νέου επαγγέλματος του Συμβούλου για την ε, χρήση αυτών των τεχνολογιών. Ένας δύο επαγγελματικό κλάδος. Τέλος, η υποστήριξη απασχόλησης. Οι βοηθητικές συσκευές για άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο, δηλαδή ε, θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση των ήδη φυστάμενων τέτοιων ε, μηχανημάτων και θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους εκ μέρους των ατόμων με αναπηρίες. Οι επαγγελματίες εδώ θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο συμβουλεύοντας τον εργοδότη για το πώς ε, μπορεί να προβεί σε μια καλή προσαρμογή προκειμένου να υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρίες στο χώρο της εργασίας. Επίσης να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση καθώς και μια, να υπάρξει μια καλή πρόσβαση στη χρηματοδότηση αυτών των ε, υποστηρικτικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρίες. Βεβαίως υπάρχουν τρομερά ελλείμματα στις ε, κοινωνίες μας και εδώ η νομοθεσία δεν μπορεί να ε, πειράσει άμεσα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της συνειδητότητας, της επίγνωσης σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και ανάγκη να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ώστε να αποφευθεί ο στιγματισμός και να προαχθεί η αποδοχή αυτών των ατόμων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μιχάλη Κρητικό. Ευχαριστώ. Mm. Βασιστήκαμε για αυτή τη μελέτη ε, στην αρχή ότι θα πρέπει να έχουμε και κάποιες νομικές και κοινωνικοηθικές διαστάσει σε σχέση με αυτά τα τεχνολογικά βοηθήματα. Έγινε εσωτερικά στη ΣΤΟΑ η μελέτη. Ποιες βασικές νομικές προκλήσεις εντοπίσαμε ε, όταν ε, κοιτάζουμε και εξετάζουμε αυτά τα βοηθήματα από ε, νομοθετικής πλευράς. Πώς ακριβώς μπορούμε ε, αυτές τις ειδικέ ανάγκες να τις εντάξουμε, ε, επειδή είναι και οριζόντιο θέμα, στην ε, αρμοδιότητα, στο φάσμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα μεικτής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Επίσης, υπάρχει νομοθετικός κατακαιρματισμός σε σχέση με τις απαιτήσει για την προσπλασιμότητα και τις προδιαγραφές στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με για τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ε, ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Ε, δεν υπάρχει οριζόντιο ε, κοινό αποδεκτό ορισμό των ειδικών αναγκών. Σε δευτερογενή νομοθεσία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, όμω σε οριζόντιο επίπεδο δεν υπάρχει κάποιο ορισμό που να γίνεται ευρέω αποδεκτό. Επίση, ευθύνη για τι ζημιέ που μπορούν να προκαλέσουν αυτόνομα τέτοια βοηθήματα που χρησιμοποιούν αυτέ τι μεθοδολογίε που περιγράψαμε και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στους χρήστες ή σε τρίτους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι ισχύει στο θέμα της ευθύνης για, τις, για τα αυτόνομα αυτά βοηθήματα. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τις νομικές διατάξεις που υπάρχουν ε, τα βοηθήματα που γίνονται αυτόνομα μηχανήματα ε, ε, οδηγούν σε σώρευση δεδομένων, μεγάλων δεδομένων που σχετίζονται με την προσωπική ιδιωτική ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή των χρηστών αυτών των ε, μηχανημάτων ε, και βάσει των οδηγιών για την ε, ίση μεταχείριση φυσικά απαγορεύεται οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε σχέση κατά κάποιο τόμο με ειδικέ ανάγκες. Προς το παρόν δεν υπάρχει όμως σχετική διάταξη μέσα σε αυτές τις οδηγίες από γνωρίζουμε. Πέραν από αυτές τι προκλήσεις, τις νομικές προκλήσεις υπάρχουν και ιδεολογικού χαρακτήρα ε, προκλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το νομικό πλαίσιο και σχετίζονται με το σεβασμό και την προστασία των βασικών θεμελιωδών διοντολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις, σχετίζονται με την αυτονομία αυτού του ατόμου που μπορεί να υπονομευθεί από αυτά τα βοηθήματα και το ίδιο και για το ναυτοπροσδιορισμό ε, ως προς την ε, πρόσβαση πληροφορίε ε, ε, και ε, την ανεξαρτησία του, δημιουργώντας νέες μορφές αποξένωσης και εγκατάλειψης. Επίσης, οδηγούν σε εξουσιοδότηση απώλεια ε, ε, ελέγχου, ε, εξουσιοδότηση άλλων, τη, απώλεια λογοδοσίας και κοινωνικής συμμόρφωσης όταν μιλάμε για την καθολική, παραδείγματος χάρη, οικουμενική προσπελασιμότητα και αποδοχή ή για τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Ε, οι αυτά τα μηχανήματα είναι πάρα πολύ ακριβά ε, και η διαθεσιμότητα στα 28 κράτη-μέλη είναι ούτως ή άλλως μεγάλη πρόκληση. Τώρα όταν, ε, όταν ε, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα μηχανήματα, μειώνεται φυσικά η ανθρώπινη επαφή ε, και ο αριθμός ε, αυτών που περιθάλπουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν είναι, είναι δυσδιάκριτη πλέον η γραμμή ανάμεσα στην στην ε, ε, βοήθεια προς αυτόν το άτομο με τις ειδικέ ανάγκες και την ενίσχυση κάποιων ε, δυνατοτήτων που έχει για, για τις καθημερινές δραστηριότητες. Επιστιγματισμός σε σχέση αυτών των ατόμων λόγω της χρήσης αυτών των μηχανημάτων και θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα μηχανήματα και να συνοδεύουν απλώς την περίθαλψη που παρέχεται από ανθρώπινα δυναμικό. Είναι λοιπόν ε, πολύ ευρύ το φάσμα των προκλήσεων νομικών και διοντολογικών. Πώ θα προχωρήσουμε. Μία σύσταση που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε την προσφυγασιμότητα. είναι υποχρέωση ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση να βρούμε ε, καινοτόμου τρόπου ε, ώστε να είναι σε σε διαθέσιμα αυτά τα ε, υποβοηθητικά μηχανήματα και οι τεχνολογίες, κυρίως σε σχέση με τα ρομπότ, ε, ούτως ώστε τα ιατρικά ρομπότ, οι ρομπότ περίθαλψης να μπορούν να αγοραστούν ε, σε προσιτές τιμές από αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο, αλλά δεν έχουν απαραίτητα την οικονομική ικανότητα να τα αποκτήσουν. Επίσης, privacy by design online. Όπως σας είπα, αυτό είναι πρόκληση για την προστασία των ε, τεχνολογικών δεδομένων. Δηλαδή, θα πρέπει ο σχεδιασμός να ε, περιστρέφεται γύρω από αυτή τη βασική αρχή της προστασίας της ιδιωτικότητας. Ε, από την αρχή του κύκλου ζωής, δηλαδή της, του τεχνολογικού βοηθήματος, θα πρέπει να λαμβάνει αυτή η αρχή υπόψη επίσης, να είναι μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες και δίκαιη διαδικασία ε, σε σχέση με την πρόσβαση στις πληροφορίες που πρέπει να θεωρείται και ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα ε, η απόκτηση ελέγχου και διατήρηση ελέγχου αυτών των ατόμων σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών βοηθημάτων ε, διότι υπάρχει το δυναμικό σε πολλά τέτοια βοηθήματα να γίνονται αυτόνομα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας ούτως ώστε να, διατηρεί τον έλεγχο και να λαμβάνει τις αποφάσεις ο χρήστη της. Ε, δομές επίσης ε, ε, οπτικές για τα διοντολογικά ζητήματα. Ε, για ε, τις ειδικές ανάγκες για τη χρήση υποβοηθητικών τεχνολογιών ε, δεν είναι πολύ συνηθισμένες αυτές οι δομές. Πρέπει να αναρωτηθούμε όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε έρθει τις δομές. Επίσης, δομή ταξινόμησης για τα υποβοηθητικά μηχανήματα θα μπορούσαμε να το λάβουμε υπόψη, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίσουμε ώστε η ανθρώπινη περίθαλψη να μην αντικατασταθεί γιατί εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη σε όλα τα κράτη-μέλη και υποβοηθητικά χρησιμοποιούνται αυτά τα βοηθητικά μηχανήματα μόνο. Ε, ε, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ε, το προσωπικό που παρέχει την περίθαψη και οι χρήστες να είναι η βασική δικαιούχοι των υπηρεσιών και να μην επικρατήσει αυτός ο ρόλος των μηχανημάτων. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας, άμα έχετε και ερωτήσεις. Ευχαριστώ για το ΕΛΚ. Ούτε ο κύριος Μπέκ, ούτε ο κύριος Κάζερ είναι εδώ. Κανείς δεν είναι. Γιαννιές από το σοσιαλιστές. Έλα, έλα εδώ. Bedankt. Excuse me, thank you for... Αχ, συγχωρήστε με και σας ευχαριστούμε για αυτή την τόσο πλήρη παρουσίαση. πάρα πολύ ενδιαφέρομαι για αυτά τα οποία είπατε και έχω κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά αυτό το οποίο μας αναπτύξατε, δηλαδή όσον αφορά το πόσο κοστίζουν τελικά, πόσο προσιτά είναι όλα αυτά τα εργαλεία, τα μέσα. Επομένως, υπάρχει και θέμα στην απασχόληση. Σε σχέση με το κόστος λοιπόν αυτών των συσκευών, θα έπρεπε να πληρώνει ο εργοδότης αυτός, θα έπρεπε να είναι ο υπεύθυνος και τι γίνεται με τους αναπήρους που δεν έχουν σταθερή απασχόληση ή τι γίνεται για εκείνου που ακόμα κάτι σπουδάζουν και δεν έχουν βρει ακόμα δουλειά. Οπότε πια δεν είναι θέμα εργοδότη, αλλά θέμα κοινωνίας. Για κοιτάξτε λίγο αυτό. Γιατί σε συνέχεια των όσων μας είπατε. Τι δυνατότητες άλλες υπάρχουν. Αν δηλαδή κανένας μπει στην αγορά απασχόλησης έχει πιο εύκολη τη λύση παρά προηγουμένως για να χρησιμοποιήσει αυτές τις υποβοηθητικές νέες τεχνολογίες και τελικά να μπορούν οι άνθρωποι να ε, συμμετάσχουν πλήρως στην ε, αγορά απασχόλησης. Επίσης, Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι αφετηρία για μια συζήτηση όσον αφορά την εταιρική ευθύνη και των εταιριών που δεν απασχολούν αναπήρως. Κάνει πιο εύκολη πως την απασχόλησε. Και έτσι έχουμε φετιρία από μέρους για αυτή την εταιρική ευθύνη και την απασχολησιμότητα πλέον αυτών των εταιριών. Τι θα μπορούσε να προβλέπετε κάποια ποσόστοση για ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία. Merci. Pour ECR, euh, e euh, Madame Stevens, éventuellement. Λύση, κυρία Stevens. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Να ευχαριστήσουμε τους ε, δύο εισηγητές. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα το μας είπαν και ε, διάβασα την έκθεση. Οπότε θα πρέπει τώρα να σας πω κάτι όσον αφορά κάποια ηθικά ζητήματα και νομικά ζητήματα τα οποία αναδύονται, τα οποία μας τα αναφέρατε και εσείς είναι πολύ σημαντικό, όπως πρώτα-πρώτα το θέμα της ασφάλειας, safety. Γιατί ε, αυτή τη βδομάδα είχαμε ένα ατύχημα με ένα από αυτά τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ε, είναι ακριβώς ζήτημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των μηχανών, των συσκευών. Αν θεωρήσουμε ότι αυτού του είδους οι μηχανές και τα μηχανήματα είναι υποβοηθητικά ή είναι ασφαλή για τους αναπήρους που τα χρησιμοποιούν αλλιώς, τότε φυσικά τα πράγματα που πάρουν στραβόδρομο Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά τους ε, ανθρώπους με κάποια αναπηρία, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο σε σχέση με αυτές τις προβλητικές συσκευέ. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό και με απασχολεί. Ποιος κρίνει πώς πρέπει να γίνεται η χρήση αυτών των τεχνολογιών. Αποφασίζουν οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρίες ή αυτοί που κάθονται σε ένα εργαστήριο και λένε «Α, πολύ καλή ιδέα αυτή για κάποιον ανάπηρο. Θα τους αρέσει πάρα πολύ αυτή μας η η εφεύρεση. Επομένως, θα πρέπει πρώτα πρώτα κανείς να βλέπει τα πράγματα από πλευρά των Χριστών και να ε, δούμε επίσης και το θέμα το ότι αυτό αποτελεί πίεση από πλευράς κοινωνίας γιατί η κοινωνία φέρνει τον ε, ανάπηρο των στριμώχνων στη γωνία και του λέει πρέπει να τα χρησιμοποιείς αυτά αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, να το δούμε από την πλευρά των Χριστών και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη, τη, γνώμη των ε, αναπήρων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν και αυτοί στο σχεδιασμό, ότι είναι που λέει ο λόγος μέσα στο εργαστήριο του σχεδιασμού. Ε, και αυτό δεν το κάνει καμία υποβοηθητική ε, τεχνολογία. Είναι δική μας κοινωνική ευθύνη. Δεν μπορεί κανένα απλώ να είναι τεχνοκράτη και να πει Μπαπ, τόλισε το πρόβλημα. Τέλειωσε. Βέβαια και κατοίκον για να μην χρησιμοποιούν τεχνολογίες. τεχνολογίε. Πολλέ φορέ δεν έχουν ε, αυτονομία και χρειάζονται την υποθετική τεχνολογία. Όμω να μην είναι δικαιολογία, πρόφαση όλα αυτά, ούτω ώστε να μην εντάσσουμε στην κοινωνία ε, τους ε, αναπήρους. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει προσβασιμότητα και στην κοινωνία. Θα πρέπει να ε, τους βοηθούμε στη μεταφορά, θα πρέπει να τους βοηθούμε να πάνε στη δουλειά τους και να μην εστιαζόμαστε μόνο στο θέμα της βοήθειας μέσα στο σπίτι. πρέπει να βοηθάμε στην ένταξη αυτών των ανθρώπων σε κάθε κοινωνικό επίπεδο και στην ε, ψυχαγωγία και στη δουλειά. Άρα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι μια λύση η υποβετική τεχνολογία, αλλά δεν τελειώνει η ιστορία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στη στάση της κοινωνίας. Οπότε και γι' αυτό συμφωνώ με τα όσα σχετικά μας είπατε. Τώρα, όσο αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου, ε, εντάξει, είναι θέμα των ίδιων των ε, αναπήρων να προστατεύουν, να είναι κάτοχοι των δεδομένων τους και να ερωτώνται εάν ε, μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε. Να μην απευθυνόμαστε σε έναν γιατρό, σε έναν επαγγελματία. Εντάξει, αυτοί να συμμετάσχουν, αλλά τελικά ο ίδιος ο ανάπηρος να είναι ο κάτοχος, ο κύριος ε, των σχετικών δεδομένων. Και αυτό αφορά και τι ασφαλιστικές εταιρείε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν εκείνες. Ε, τώρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση βέβαια. Να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρεών, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε σχέση με το ποιος πληρώνει για αυτά τα υποβευτικά μηχανήματα. Είναι Πάμε θέμα κοινωνικής ευθύνης, θέμα κρατικής ευθύνης, να εξασφαλίσουμε ότι οι ανάπηροι έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή, να τους βοηθήσουμε, ώστε να έχουν αυτονομία στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλον από άλλη πολιτική ομάδα. Ούτε για τους πρασίνους. ζήτη κανείς το λόγο. Η FTD κανείς. Ντομινίκ Μαρτέν. Όχι, δεν θέλετε το ρόλο. Αλλά ο κύριος Φουντούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με σύνδρομο Down και έχω προσωπικούς λόγους να έχω ένα αυξημένο ενδιαφέρον σαν γονέας μιας κόρης με σύνδρομο Down για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες τόσο τα άτομα με νοητική στέρηση, αλλά και άλλες μορφές αναπηρίες όπως κινητικές, οπτικές, ακουστικές κλπ. Η μελέτη, την οποία θα διαβάσω με μεγάλη προσοχή, δυστυχώς περιορίζεται μόνο στα θα και όχι στο πώς. Θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να θεωρείτε κλπ. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά μπορώ να έχω ήδη αντίληψη για το τι συμβαίνει στη χώρα μου την Ελλάδα. Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες είναι το πρώτο και βασικό βήμα για την εξέλιξη της πορείας της ζωής τους και για την ένταξη στην αγορά εργασίας, που είναι και το ζητούμενο. Στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρίες έχουν υποστεί όλα τα δεινά της οικονομικής κρίσης. Παράλληλη στήριξη δεν υπάρχει για τα άτομα με αυτισμό στα περισσότερα δημόσια σχολεία. Ακόμα και για τα εργαστήρια στα ειδικά σχολεία δεν θα μιλήσω για το απλήρωτο εκπαιδευτικό προσωπικό ή την έλλειψη θέρμανσης. Θα επισημάνω όμως ότι δεν υπάρχουν ούτε υλικά για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικέ ικανότητε. Οι υποστηρικτικέ τεχνολογίε για τα άτομα με αναπηρίε μπορώ να πω πω είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δυστυχώ στην πράξη είναι απλά ευχολόγια και η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή που μα διαψεύδει. Ευχαριστώ. Merci. Euh, euh, la parole à nos collègues, euh, je sais pas, monsieur. Ευχαριστούμε τον ε, λόγο στους δύο εισηγητές μας για να απαντήσουν στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Κύριος Κρητικός, η κυρία Μάγια. Thank you so much for the interesting... Uh, Ευχαριστούμε, λέει η κυρία Μάγια, για όσα ακούσαμε για την μελέτη αυτή και έχουμε διάφορα σημεία που έφυξαν οι διάφορες ερωτήσεις. Αρχή, αρχή, μα είπατε για τι ποσοστώσει. Ναι, σε κάποιε χώρε έχουμε ποσοστώσει. Και ένα τμήμα τη μελέτη που κάνουμε με στόχο να υπάρξει σχετική νομοθεσία. Κάτσαμε και καταγράψαμε λοιπόν τι προβλέπουν νομοθεσίε σε όλη την ε, Ευρώπη και καταλήξαμε σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, Γερμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σουηδία και είπαμε ότι αυτές οι χώρες εκπροσωπούν άλλες περιοχές της Ευρώπης οπότε και συνειδητοποίησαμε ρετώντα αυτέ τι τέσσερι ε, διαφορετικέ περιπτώσει τι γίνεται με τι ποσοστώσει. ότι σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτικές οι ποσοστώσεις. Αλλά στην ε, Γερμανία, Φερρυπίν, αφορούν ε, και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτές τις ποσοστώσεις του επιβάλλεται πρόστιμο και στην Πορτογαλία υπάρχουν ε, ποσοστώσεις, αλλά μόνο για το δημόσιο. Οπότε και εδώ είναι μια δυσκολία, διότι είναι θετικό το ότι υπάρχουν ε, ποσοστώσεις. Το θέμα είναι όμως πώς το εποπτεύει κανείς αυτό. Ούτε έχουμε αρκετά στοιχεία για το τι γίνεται. Τι γίνεται με τους αναπήρους. Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα και στοιχεία. Βεβαίω, έχουμε και κάποια αξιόλογα παραδείγματα στην Πορτογαλία και τη Γερμανία. Εάν οι εργοδότες αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει σημαντική, σοβαρή προσπάθεια απασχόλησης και ότι έχουν εξασφαλίσει κατάλληλους χώρους, τότε αμείβονται. Υπάρχουν δηλαδή οικονομικά κίνητρα. Λαμβάνουν κάποιο είδους οικονομική ενίσχυση. Και επίσης δικαιούνται οι εταιρείε να το προβάλλουν αυτό. Ότι δηλαδή απασχολούν ε, πρόσωπα με αναπηρίες και το ότι έχουν ε, αναλάβει τις κοινωνικές τους ευθύνες κλπ. Κύριε θέλετε κάτι να προσθέσετε. Μετά, μετά. Άλλο ενδιαφέρον αναφέρθηκε το θέμα του ελέγχου των υποβλητικών τεχνολογιών. Και επίσης όσον αφορά την προσέγγιση επί τη βάση του χρήστη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις υποβοηθητικές, αφορά όλες τις τεχνολογίες. Συνήθως η βιομηχανία προωθεί την τεχνολογία σε διάφορους τομείς και εν προκειμένου. Οπότε θα πρέπει ο χρήστης να μην βρίσκεται απ' έξω από τις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης τεχνολογίας. Θα πρέπει να έχουν λόγο και οι χρήστες. Τι χρειάζονται από την τεχνολογία. τι θέλουν ακριβώς να κάνουν και να τους βοηθήσει αυτό η τεχνολογία. Δεν είναι θέμα του να επισκευάσει κανείς κάτι που δεν πάει καλά στο σώμα του το θέμα, είναι οι ανάπηροι άνθρωποι να παρακάψουν τους φραγμούς τους κοινωνικούς που έχουν μπροστά τους. Οπότε, θα πρέπει να τους συμπεριλάβουμε τους χρήστες, τους ανάπηρους στην υπόθεση αυτή. Να, ποια είναι η γενοτομία στην ε, υπόθεση της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών. Φυσικά φραγμοί υπάρχουν και προέρχονται από την κοινωνία. Το πώς θα μπουν στα κτίρια, πώς μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πάρκο. Οπότε, για παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποια κυρία έχει ένα μωρό σε ένα καρότσι, εάν έχει σκαλιά, πώς θα σηκώσει το καρότσι να ανέβει τα σκαλιά για να πάει με το μωρό στο πάρκο. Μα, το ίδιο συμβαίνει και με άνθρωπο με αναπηρία. Τα εμπόδια από την κοινωνία τα οποία πρέπει να παρακαμφθούν. Και στο χώρο εργασία ισχύει αυτό. Σα είπα κάποια παραδείγματα στην παρουσίαση. Κάποια απλά πραγματάκια που θα μπορούσε να κάνει ο εργοδότη και πολλές φορές δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Μα είπε ένα από τους εμπειρογνώμονε ότι έχει στον υπολογιστή του κάποιες βοηθητικές τεχνολογίε, Αλλά δεν χρειάζεται να πάρει τον υπολογιστή αυτό στη δουλειά, γιατί στη δουλειά έχει ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή είναι μια εφαρμογή που μεγαλώνει την οθόνη, να διαβάσει πιο εύκολα. Και άλλε ε, ε, μια άλλη που μεταφράζει σε εικόνα τη λέξη, οπότε μπορεί να καταλάβει καλύτερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν δεν υπάρχουν αρκετέ πληροφορίες δεν υπάρχει προσβασιμότητα των αναπήρων στον χώρο τη δουλειά. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να συνειδητοποιηθούν και φυσικά να δοθούν και κίνητρα. Ε, αν κανείς να λαμβάνει τις ευθύνες του, τότε να επιβάλλονται αυτές. Κάτι σαν πρόστιμο, κάτι που πραγματικά να υποχρεώνει τις ε, εταιρείε να χρησιμοποιούν υποβεστικές τεχνολογίες. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της ε, κατοχής, της κυριότητας των ε, δεδομένων. Φυσικά και αυτή ανήκει στον χρήστη. Αλλά ένας ειδικό, ένας εμπειρογνώμας μας είπε ότι όταν έχουμε τέτοιες καινούργιες τεχνολογίες, όπως το, αυτό που πρέπει να πάει στον χώρο της δουλειάς, θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται εκτός στο δρόμο όταν κάποιος, ας το πούμε, εξασκείται ε, σε αυτή την ε, ε, κατοικόνα πραγματικότητα, την εικονική πραγματικότητα, στο πώς θα αντιδράσει στη μηχανή, τα, σχετικά με τις μηχανές. Απαιτούνται δεδομένα όχι μόνο από το χρήστη, αλλά και από το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς τους κοινωνικούς κανόνες για τα δεδομένα και κατά πόσο οι άλλοι θέλουν τα δεδομένα τους να τα μοιράζονται με τον χρήστη με τέτοιες τεχνολογίες. Γιατί σε τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να συλλέξει δεδομένα αλλωνών ο χρήστης. Άρα αυτό αξίζει να μας προβληματίσει περισσότερο. Α, αυτό το τελευταίο που άκουσα από τον κύριο από την Ελλάδα, ναι. Εγώ είμαι Πορτογαλέζα έχουμε παρόμοια κατάσταση και υπάρχει παρόμοια δυσκολία. Όταν κάποια χώρα έχει οικονομικές δυσχέρειες, ε, δύσκολο είναι να κάνουμε αυτό το οποίο είπατε. Αλλά κάποια πράγματα ε, τα μάθαμε από αυτή τη μελέτη μας, έδωσε ιδέες και προσπαθούμε σε τέτοιες μελέτες να δούμε ποιες είναι οι άρεθες πρακτικές παραδείγματα προς μίμηση. Τι κάνουν δηλαδή άλλες χώρες για να τα πάρουμε να τα κάνουμε και στη δική μας. Να, ένα καλό παράδειγμα από την Πορτογαλία. Έχουμε τα ειδικά σχολεία. Κλείσανε. Δεν έχουμε τώρα. Οπότε όλοι οι μαθητές από εκεί εντάχθηκαν στα συνήθη σχολεία. Να, ποια είναι η παιδεία χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης και κάτι άλλο μπορεί κάνει να εμπνευστεί από την Πορτογαλία, σχολεία ή πανεπιστήμια που δεν ήταν υποχρεωμένα να δώσουν υποβεθυντικές τεχνολογίες στους μαθητές και φοιτητές. Δηλαδή υπήρχε η ιδέα αλλά δεν δόθηκε η σωστή συνέχεια. Να, κάτι που είναι στην Πορτογαλία και θα μπορούσε αν το αντιμετωπίσει και αλλού. Στο άλλο άκρο είναι η Γερμανία. Υπάρχουν ακόμα ειδικά σχολεία. Και σχολεία και πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να παράσχουν την υποβευτική τεχνολογία. Επομένως, εντάξει, δεν είναι το παν το χρήμα. Και έχουμε πολλές Τέτοιε τεχνολογίες που κυκλοφορούν στην αγορά. Θα πρέπει όμως να τις μάθουμε καλύτερα, θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή των υπαρχουσών τεχνολογιών και αντί να ξοδεύουμε τα λεφτά μας στην υψηλή περίπλοκη τεχνολογία που θα είναι μόνο σε λίγους προσβάσιμη κοιτάξουμε αυτό το θέμα του κόστους. Γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες υποθετικές ε, τεχνολογίες που ονομάζονται ιατρικές συσκευές και έχουν σχέση και με το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, εάν κάποια τεχνολογία είναι θέμα ε, ιατρικής, μα τότε έχει περάσει από χίλιους ελέγχους για να χαρακτηριστεί ιατρικό εργαλείο, ιατρική μέθοδος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είμαστε εντάξει από πλευράς ασφαλείας. Δεν έχουμε το πρόβλημα. Επίσης και κάτι άλλο που βρήκαμε μπροστά μας στη μελέτη είναι το αν θα πρέπει όλες οι υποθετικές τεχνολογίες να χαρακτηριστούν ε, ιατρικά μέσα. Ούτως ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα από όλο τον κόσμο. και σαν πρόταση είδαμε το ότι ένα πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία κρατάει πάρα πολύ χρόνο για να χαρακτηριστεί μια συσκευή ιατρική. Οπότε η βιομηχανία δεν έχει κίνητρο να προωθήσει τέτοιες συσκευές που θα χαρακτηριστούν κάποια στιγμή ιατρικές. Νομίζω ότι πρέπει να βάλω εδώ τελεία. Ναι, ναι, ναι, ναι πιεζόμαστε από τον χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη που μακρηγόρησε, λέει κύριε Μάγια, αλλά είχαμε τόσα θέματα. Ναι, ναι, ναι, αλλά τα είπατε όλα και νομίζω ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Άρα, σημαντικό το ότι μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Πάμε τώρα στις μία αυτά της μερικής διατάξεως. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 19. Εδώ Πρέπει να κάνουμε ανταλλαγή απόψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε κάποια έξι πιλωτικά προγράμματα. Οπότε θέσαμε αμέσως να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σούκοβα. Ε, αναπληρώτρια διευθύντρια της ε, Γενικής Διεθνής για την Απασχόληση. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας κάνω παρουσίαση τριών προγραμμάτων στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόληση και είμαστε... Η αρμόδια αρχή για την έγκριση των οικονομικών εντολών. Ε, λοιπόν, στις 27 Φεβρουαρίου 2018 ήταν η, η έγκριση του προγράμματος. Βλέπετε τις λεπτομέρειες για τους στόχους και για την φάση εφαρμογής για τα προγράμματα. Για και για τα προηγούμενα χρόνια και για τα προγράμματα που θα τρέψουν το 2018. Επίσης, ενδεικτικά ε, δίνεται και μία πρόβλεψη για το χρονοδιάγραμμα για τα βασικά βήματα. Και ε, για όλα αυτά τα στοιχεία θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Θα καταρτιστεί και δεύτερη έκθεση με την οικονομική δήλωση που θα διαβαστεί στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019. Το Μάιο θα τη λάβετε. Λοιπόν, ε, έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της αρμοδιότητας ε, της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επασχόλησης και δύο προπαρασκευαστικές ε, δράσεις. Η, τα, τα δελτία υπηρεσιών, service vouchers και η οικιακή βοηθή, τα, επίσης το, η εγγύηση για τα παιδιά. Το πρώτο πρόγραμμα, να δούμε με τη σειρά, για τους υγειακούς βοηθούς και για τα προγράμματα με τα δελτία παροχής οικιακών υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα για να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία και για να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για αυτούς που προτείνουν, παρέχουν αυτές τις ε, προσωπικές υπηρεσίες και οικιακές υπηρεσίες. 700.000 ε, ευρώ για είναι το ποσό και δύο βασικοί στόχοι. Όπως είπαμε, τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τέτοια καθεστώτα για τα δελτία υπηρεσιών και να ενισχύσουμε ε, τον κοινωνικό διάλογο σε αυτό το τομέα. Συμβουλές, τεχνική αρρωγή και ε, διάφορες ε, Συστάσει και κατευθυντήρια σε γραμμέ, προσαρμοσμένες ανάγκε των κρατών μελών για την ενίσχυση αυτού του τομέα των οικιακών υπηρεσιών. Επίση, θα υποστηρίξουμε την ανταλλαγή ε, βελτίστων πρακτικών ανάμεσα στις, ε, ε, στους ΧΙΤΑ, στις εθνικές αρμόδιες αρχές, στις οργανώσεις οικιακών βοηθών και προσωπικού περίθαλψης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ε, να ε, ε, διάδοση των πληροφοριών για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, τους ώστε να αναγνωριστεί αυτό το επάγγελμα και όπως είπαμε να ενισχύσουμε και τον κοινωνικό διάλογο σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, ε, για τον τομέα αυτό να σας ε, θυμίσω ότι στην από δύο ε, τμήματα. Ε, οι υπηρεσίες σχετίζονται με την περίθαλψη ε, κατοίκων παρέχονται για την περίθαλψη παιδιών, ηλικιωμένων, αρρώστων, ατόμων με ειδικέ ανάγκες και Δεύτερο, δεύτερη κατηγορία, οι υπηρεσίες οικιακές, ε, καθαρισμός, ε, σιδέρωμα, φροντίδα του κήπου, ε, συντήρηση κτλ. Επιδιορθώσεις. Και εδώ έχουμε δύο υποκατηγορίες, τους παρόχους υπηρεσιών και τα μέλη της οικογένειας για τα οποία δουλεύουν. Μπορούμε να δείξουμε κάτι, όχι. Η βασική ενδιαφέρον είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τους εργαζομένους σε αυτό το τομέα, θεακές υπηρεσίες, ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και η εκπρόσωπη των εργαζομένων αυτό το τομέα, Global Europe, ε, Συνδικάτο Global Union Europe. Αυτή θα είναι η βασική εταίρη μας για την εφαρμογή αυτών των ε, πιλωτικών προγραμμάτων. Τι, ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος ε, και ε, του ομίλου που θα επιλεχθεί και πρέπει να αναπτύξει τουλάχιστον τις εξής δραστηριότητες. Πρώτον, τα κράτη-μέλη που είναι πιο προχωρημένα σε σχέση με την ε, ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών θα οργανώσουν τη, ε, θα οργανωθούν γύρω από δύο βασικές δραστηριότητες, συλλογή ευελίξεων πρακτικών για την ε, ανάπτυξη επίσημης απασχόληση σε αυτόν τον τομέα και ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου για τους οικιακούς βοηθούς. Ε, υπάρχουν και κράτη-μέλη όπου Αυτέ οι υπηρεσίε περίθαλψη και οι οικιακέ υπηρεσίε δεν είναι τόσο ανεπτυγμένε, οπότε θα επικεντρωθούν τα κράτη-μέλη στην διάδοση καλών πρακτικών και την τεχνική αρρωγή και οι δραστηριότητες που προβλέπουμε να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οργάνωση ευρωπαϊκής διάσκεψης, Οργάνωση και τροφοδότηση μια ιστοσελίδα με τι καλέ πρακτικέ, ε, διαθέσιμε πληροφορίε μέσα τη ιστοσελίδα και τεχνική αρρωγή των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων όταν ε, ε, θεσπίσουν αυτό το σύστημα δελτίων υπηρεσιών και ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δώσει επιδοτήσεις για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και ε, γίνεται πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Ε, αρχίζει τις επόμενες εβδομάδες. Θα επιλεχθεί μια, ένας όμιλος και τις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιευθεί η υποβολή. Η διορία για την υποβολή προσφορών θα είναι τέλη Ιουνίου ε, και θα προβλέπεται ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχουμε υπογράψει για την επιδότηση για να αρχίσει και η εφαρμογή του πιλωτικού. Δεύτερη, προπαρασκευαστική δράση, εγγύηση για τα παιδιά. Είναι στο δεύτερο έτος εφαρμογής ήδη το αρχικό πρόγραμμα ασχολήθηκε με τη χαρτογράφηση της ε, κατάστασης ε, για την αποτελεσματική ε, προστασία και σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, ανάλυση του των όρων της προσθέμενης αξίας και του εφικτού αυτής της εγγύησης για τα παιδιά και Μιλάμε για παιδιά που ζουν σε ασφαλέ πέσει θέμα, θύματα εμπορίας ή έχουν ειδικέ ανάγκες. Η σε οργανισμους εχουν πεσει θεμα θυματα εμποριας η εχουν ειδικε αναγκες η προετοιμασια της σε δράση, λοιπόν προϋποθέτει η εφαρμογή ενός πλαισίου ε, για, να, για το, το καθεστώς αυτό, για τα αποτελέσματα της πρώτης πρωτοπαρασκευαστικής δράσης, του πρώτου σταδίου δηλαδή, αν θέλετε, της πρωτοπαρασκευαστικής δράσης, θα πρέπει να ερευνήσουμε ε, σε ποιο βαθμό τα πορίσματα της πρώτης δράσης ε, θα μπορέσουν να διευρυνθούν για να καλύψουν αυτές τις κατηγορίες παιδιών ε, ή δυνατόν σε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εγγύηση για τα παιδιά, λοιπόν, ε, μελέτη ε, ε ε, ε, λίγη προθεσμία τον Απρίλιο του 2018 σε ένα μήνα και ε, προετοιμάζουμε και την οικονομική απόφαση για την επέκταση, για το δεύτερο δηλαδή στάδιο της προπαρασκευαστικής δράσης θα χρηματοδοτηθεί από το προϋπολογισμό το 2018. Η εκπόνηση της μελέτης, για να δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες αν μου επιτρέπετε, ε, στοχεύει την συλλογή γνώσεων για την προπαρασκευαστική δράση, ε, συλλογή πραγματογνωμοσύνης από τους ενδιαφερομένους μέσω ειδική διαβούλευσης, ε, input από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δημοσιολαβητών για τα Παιδιά, για να συζητήσουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του Συμβουλίου η επέκταση του προγράμματος που είπαμε θα χρηματοδοτηθεί από τον προπολογισμό του 2018 θα βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και θα καταδείξει τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της πρώτης δράσης και θα μας θα προτείνει συγκεκριμένα βήματα για τη δεύτερη φάση. Επίσης, ε, προπαρασκευαστική δράση, reactivate λέγεται, είναι μια δράση που συνδέεται με μελέτη αποτελεσματικότητας ενός ε, Ευρωπαϊκού Συστήματος Κινητικότητας για ανέργους ε, άνω των 35 ετών για τους μακροχρόνια ανέργους κυρίως για να βρουν ε, μια θέση εργασίας ή τουλάχιστον ευκαιρίες για μαθητεία, παραδείγματος εργασία ε, η προσπάθεια αλλο κράτο μέλο, να ενισχυθει η προσπαθεια σωμάτωσή του στην αγορά εργασία και επίσης να βελτιωθούν οι συνθήκες για την εξέβραση εργασία για να μπορέσουν να ασκούν την ελευθερία ε, μετακίνησης ως Ευρωπαίοι πολίτες και για να καλύψουμε τις ελλείψεις ε, που ε, υπάρχουν στις αγορές εργασίας σε διαφόρων κρατών μελών, ε, να γίνει καλύτερη αντιστοίχηση αυτών που ψάχνουν δουλειά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Το 2016 είδατε δαπανήθηκαν 3 εκατομμύρια, 2,5 το 2017 και άλλα πέντε ε, στο προϋπολογισμό του 2018. Συνολικός προϋπολογισμός, δηλαδή η χρηματοδότηση του προγράμματος ε, θα ανέλθει στα 10 εκατομμύρια και μισό. Τα μέτρα υποστήριξη ε, προς τους δικαιούχους του προγράμματος θα είναι πολλά και διαφορετικά ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ε, βοήθεια για να κάνουν συνεντεύξεις στην Αλλοδαπή ή ε, γλωσσική ε, γλωσσικά μαθήματα για όσους θέλουν να μετικήσουν ε, και βοήθεια για αυτές τις ε, μαθητείες που ενδεχομένως βρουν ή τα στάσει σε κάποια άλλα κράτη-μέλη που βοήθησε προς μικρές νομικές οντότητες αυτοαπασχολούμενων και επιλέγουμε φυσικά την απλουστευμένη μέθοδο κοστολόγησης και προβλέπεται μεικτή χρηματοδότηση. Ε, τα προγράμματα από τρεις μήνες για μαθητεία έως έξι μήνες αν ε, πρόκειται για στάση ε, και υποστήριξη αν τελικά αποφασίσουν να μείνουν στο κράτος μέλος οι δικαιούχοι και να βρουν δουλειά. Τρίτο στάδιο για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος το 2018 εξαρτάται βέβαια και από την έγκριση τη δημοσιονομική απόφαση που είπαμε επίκειται ε, η πρόταση, η πρόσκληση μάλλον για υποβολή προσφορών θα δημοσιευθεί με το που εγκριθεί η δημοσιονομική απόφαση και ε, στο τρίτο τρίμηνο προβλέπεται έναξη του προγράμματος. Μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη φάση της προπαρασκευαστικής δράσης, απλούστευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα, τους ομίλους που μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Ε, είχαμε ε, πάρα πολύ λίγες προσφορές ε, και αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, να ενισχύσουμε δηλαδή διασυνοριακά και διαπεριφερειακά προγράμματα και γι' αυτό προτείνουμε δύο και όχι τρεις εταίροι να είναι επιλέξιμοι, για τους ομίλους πάντα μιλάμε. Ε, επίσης, ε, η οικονομική υποστήριξη για την ε, ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και για τις επιδοτήσεις Προτείνουμε 1.200 ε, ε, δράσεις υποστήριξης ε, με δεκτικό χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Αυτό το στάδιο του προγράμματος μπορεί να είναι οι υπηρεσίες ιδιωτικές ή δημόσιες, αλλά να ανήκουν κυρίως στο δίκτυο Γιούρες για την εξεύρεση απασχόλησης και πιστεύουμε ότι με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να Ε, επιταχύνουμε έτσι την κινητικότητα των ανέργων και επίσης να διευρύνουμε τις δραστηριότητες στήριξης για όσους ε, δεν μπορούν να βρουν μια κατάλληλη εργασία ως προς τα προσόντα τους στο κράτος μέλος που διαμένουν και θέλουν να μετηγήσουν την Ελλοδαπή. Αυτά, αυτά τα πιλωτικά και προπαρασκευαστικέ δράσεις είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε να συζητήσουμε το περιεχόμενο ε, των προτινόμενων μέτρων για το 2018 δηλαδή. Ευχαριστούμε. Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Η Μαρίτα Ολσκόκ που είναι η συγγήτρια όπως σας έλεγα δεν μπορεί να είναι εδώ. Η Αγνές όμως ε, θα μιλήσει από εξονόματος της Μαρίτας. Not on Marita's ε, Εκ μέρους της Μαρίτας. Γιατί να μιλήσω εκ μέρους της Μαρίτας. Θα μιλήσω σε σχέση με την προπαρασκευαστική δράση όσον αφορά την εγγύηση υγείας, για την υγεία, γιατί είναι αυτό το, το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα και συνιστά και μια προτεραιότητα για τη δική μου πολιτική ομάδα εγκρίθηκε το 2016 για τον προπολογισμό του 2017 και εφόσον υπάρξει η προκήρυξη, η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού ε, έγινε πριν από μερικούς μήνες και θα ήθελα να μάθω γιατί έγινε αυτό εφόσον εγκρίθηκε το 2016 για τον προπολογισμό του 2017 μέχρι, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε τον Απρίλιο του 2018 εσώ τουριστικοποιηθούν όλα τα προγράμματα γιατί ε, χρειάστηκε να περάσει τόσος καιρός έως ότου δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, όσον αφορά το πρώτο τμήμα της προπαρασκευαστικής ε, δράσης, πρόκειται για την εγγύηση για τα παιδιά. Ε, το πρώτο τμήμα έχει εφαρμοστεί και αν όχι, πώς μπορεί να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Και τέλος, το, έχει υποβληθεί το αίτημα να ανατεθεί η προπαρασκευαστική αυτή δράση στο Eurofound. Και το ερώτημά μου έχει ως εξής. Πώς, ε, ε, τι πιστεύετε εσείς, δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να χρησιμοποιηθεί μια πραγματογνωσύνη του Eurofound γιατί νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης και στη διαδικασία εφαρμογής. Και θα ήθελα να μας πείτε και τη δική σας άποψη για την ιδέα αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, από το Άλντε, κυρία Μάρκιν, από την Κούε, θέλει να μιλήσει κανείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και ε, όσον αφορά τις ε, λεπτομερείς ε, πληροφορίες που μας έδωσε για αυτό το πρόγραμμα πιλότος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ειδικά όσον αφορά τις κερκές βοηθούς γιατί αυτό το πρόγραμμα το προωθήσαμε τον περασμένο χρόνο και είχε πολύ καλή υποδοχή από την Επιτροπή Απασχόλησης του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή και γι' αυτό την ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι μια προτεραιότητα όσον αφορά την ομάδα μου και την δική μου εργασία προσωπικά. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο χρόνο ε, οι ομάδες των οικιακών ε, βοηθών με τις οποίες είμαστε σε επαφή στην Ισπανία ε, χάρηκαν πολύ και το είδαν σαν ένα βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίων τους ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται διαφορετικά και έχουν επίσης θετικές προσδοκίες όσον αφορά τη βελτίωση των συνθήκων εργασία. Ε, είχα κάποιες ερωτήσεις, ε, πολλές από αυτές ε, καλύφθηκαν από την αρχική σας παρουσίαση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν έχετε ξεκινήσει κάποιο διάλογο με τις χώρες μέλη και αν τι είδου αντιδράσχαν, ήταν θετική υποδοχή τους επιθυμούν να τα εφαρμόσουν για να βελτιώσουν τον κοινωνικό διάλογο. Επίσης, τα... Επίσης ε, κατά πόσο θα τεθούν στην διάθεση τα στοιχεία αυτά, ε, οι αυτές για, ε, στη διάθεση των τοπικών κυβερνήσεων ή των τοπικών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι θα προτείνουμε φέτος μια δεύτερη φάση αυτού του προγράμματος, του project, το οποίο θα έχει σαν στόχο να προωθήσει μια συγκεκριμένη πιλωτική εμπειρία, πιλωτικό πρόγραμμα ε, σε μικρή κλίμακα ενδεχομένως, σε περιφερειακό επίπεδο, ούτω ώστε να προωθήσουμε περισσότερο τις ε, συνεταιριστικές ε, ενώσεις των εργαζομένων ε, γυναικών οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιους συνεταιρισμούς να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες ούτως ώστε να το πετύχουν πιο αποτελεσματικά. Για τους πρασίνους, όχι δεν θέλετε να πάρετε το λόγο, άρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στις διάφορες ερωτήσεις που υποβλέθηκαν. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας όσον αφορά αυτό μας το πρόγραμμα και την εφαρμογή του. Και με αυτή την εγγύηση τελικά καθυστερήσαμε να αρχίσουμε. Α, σήμερα μόλις δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός. Σύμπτωση. Είδατε. Και Συζητάμε τι θα γίνει με το πιλωτικό πρόγραμμα, αν μπορεί να γίνει κομμάτι του EASY και τελικά ε, άργησε να ψηφιστεί η έγκριση του, του προγράμματος του 2017 για να δούμε το πώς θα στήσουμε αυτό το πρόγραμμα της εγγύησης για τους ανηλίκους. Ε, τελικά μας πήρε παραπάνω όπως υπολογίζαμε η προετοιμασία, να δούμε τι θα καλύπτει η πρώτη φάση και τι δεύτερη. Οπότε και πιστεύω ότι τώρα που έχει γίνει η δημοσίευση θα έχουμε τις προσφορές και θα πάμε σε μια πραγματική εφαρμογή γιατί για κάποια παιδιά σε όλα τα κρατη χρειάζονται την προστασία και χρειάζεται επίσης και πράσπιση των δικαιωμάτων τους. Μας είπατε επίσης ότι το Eurofund θα βοηθούσε. Ε, ναι, αλλά είναι το θέμα της έμεσης διαχείρισης και το ότι το πιλωτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να πάει και αυτό εκεί. Αυτό σημαίνει ότι, ότι εμείς το εφαρμόζουμε. Σύμφωνα με τις κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού επίσης θα έπρεπε να έχει οριστεί το πώς θα γίνει η υλοποίηση, πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια. Αυτό όμως δεν περιλήφθηκε στην σχετική απόφαση, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί κάποια μελέτη, κάποια ανάλυση και θα το έκαναν αυτό οι εξωτερικοί φορείς καλύτερα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες κατοίκων, είπαμε ότι πρόκειται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ούτω ώστε την αδύρωτη εργασία να την καταπολεμήσουμε και είπαμε ότι υπάρχει σχετική πλατφόρμα για την αδύρωτη εργασία οπότε και εκεί συζητούνται τα σχετικά. Ε, εκεί παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, έτυχε ευμενέστατες υποδείξεις από τα κράτη-μέλη. Ε, όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι όλα αυτά καλύπτονται επαγγελματικά και παρέχονται επαγγελματικά, αλλά και το ότι οι παρέχονται τις υπηρεσίες να είναι θωρακισμένοι, να έχουν ε, τα δικαιώματά τους όπως θέλει να τα έχει ο κάθε εργαζόμενος. Προσπαθήσαμε επίσης να επιταχύνουμε την εφαρμογή του προγράμματος και τελικά αυτό έχει σχέση και με τους στόχους του κοινωνικού πυλώνα. Δίκαιες συνθήκες για όλες τις εργασίες. Και όπως σας είπα, είμαστε σε προχωρημένο σημείο σε σχέση με τον διαγωνισμό. Και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα από φέτος. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω τελειώσαμε. Θα σας στείλω το χρονοδιάγραμμα με email. Αλλά θυμηθείτε 23 Απριλίου για διαβίβαση των ε, προτάσεων για το πιλωτικό πρόγραμμα και 29 το πρωί θα γίνει η συζήτηση ψήφιση. Δυόμιση ώρα θα αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες.